We resume the Ζητώ συγγνώμη για την καθυστέρηση. Περνάμε τώρα στην εξέταση των τροπολογιών για τη νέα ευρωπαϊκή στρατηγική για τις διεθνείς πολιτισμικές ε, σχέσεις. 313 τροπολογίες. Έγινε μια συνάντηση των σκιωδών στις 26 Απριλίου οι δύο εισηγητές συζήτησαν και συμφώνησαν για 21 συμβιβαστικές οι οποίες θα πρέπει να ψηφιστούν. Θα δώσω λοιπόν τον λόγο στον συμπρόεδρο η οποία θα διευθύνει τις ε, συζητήσεις από εδώ και πέρα. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Πρόεδρε, κυρία Πρόεδρε που μου δίνετε την ευκαιρία να πω δύο λόγια. Α, δεν λέει ο κύριος Μπροκ που πήρε το λόγο. Sorry, Mr. Brock. Ε, it is my turn. Συγγνώμη κύριε Μπροκ, αλλά ήταν η σειρά μου. Αναλαμβάνω την προεδρία της συνάντησης. Ευχαριστώ τον προηγούμενο ομιλητή και θα συνεχίσω στην ουγγρική γλώσσα. Ευχαριστώ λοιπόν για μια ακόμη φορά. Πριν δώσω το λόγο στους υπόλοιπους εισηγητές, να μου επιτρέψετε να κάνω μια μικρή εισαγωγή. Τα τελευταία χρόνια η Ευρωπαϊκή Ένωση ζει σε μια κρίση οικονομική και κοινωνική. Και υπάρχει ένα στοιχείο το οποίο ελείπηθα, αν θέλετε, από την προσπάθεια που κάνουμε για να βγούμε από την κρίση και αυτό είναι ε, ο πολιτισμός. Η δημοκρατία εξαρτάται από τον πολιτισμό. Εμείς στην Επιτροπή Πολιτισμού θεωρούμε ότι είναι πολύ σημαντικό να εμπλέξουμε τα θέματα του πολιτισμού στις συζητήσεις οι οποίες γίνονται για το ποιες πολιτικές θα ακολουθήσουμε από εδώ και πέρα. Ο πολιτισμός δίνει ουσία στη ζωή και είναι μία από τις βάσεις της κοινωνίας μας σήμερα. Ευχαριστώ τους δύο εισηγητές που προετοίμασαν μια ισχυρή πρόταση η οποία περιγράφει την αξία την οποία έχει ο πολιτισμός και εισάγει τον πολιτισμό σαν την μηχανή αν θέλετε πίσω από τις κοινέ ε, διεθνείς σχέσεις. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε, κύριε Πρόεδρε. Δεν χρειάζεται εγώ να μακρηγορήσω. Έχουμε ξανακάνει τη συζήτηση αυτή στο παρελθόν. Και δεν μπορώ να συμφωνήσω με την κυρία Μπόξορ. Τα έχουμε συμφωνήσει, τα έχουμε κανονίσει. Είδαμε τις τροπολογίες που κατατέθηκαν στις συνεδρίες των σκιωδών, εισηγητών, εξαντλητικά τις έχουμε συζητήσει και με μεγάλη υποστήριξη, αν δεν απατώμε. Στη συμβαστική τροπολογία παριθμών 2 χρειάζεται λίγη δουλειά ακόμα, γιατί δεν έχουμε προχωρήσει επαρκώς ε, δεν έχουμε βρει τον ε, επιθυμητό συμβιβασμό, πράγμα που σίγουρα θα κάνουμε στη συνέχεια, ε, για το, ιστορική κληρονομιά και πολιτιστική κληρονομιά στην Ευρώπη. Δεν έχουμε συμφωνήσει τι εμπεριέχει. Ορισμένοι θέλουν να μιλήσουν σε φιλοσοφίες και δικαιώματα από την ελληνορωμαϊκή εποχή, από την ουδεοχριστιανική σκέψη, από το διαφωτισμό και μέχρι το Ισλάμ. Ό,τι υπάρχει σήμερα στην Ευρώπη δεν σημαίνει ότι είναι και κληρονομιά της Ευρώπης. Εν πάση περιπτώσει αυτά θα τα βρούμε και είμαι πεπισμένος ότι και τις επόμενες ημέρες θα υπάρξει ένας ε, λογικός συμβιβασμός. Πρώτον για να μην πούμε τίποτα λανθασμένο και δεύτερον για να είναι όλοι ικανοποιημένοι και ευτυχείς. Για να προσθέσω και έναν άλλο φιλόσοφο, το Leibniz, Είμαστε υπέρ του ε, καλύτερου κόσμου, όλων των κόσμων. Αλλά είναι ενδιαφέρουσα άσκηση. Για την Επιτροπή Πολιτισμού, ο πολιτισμός είναι ε, αξία από μόνος του. Ενώ για την ΑΦΕΤ, την Επιτροπή Εξωτερικών, ο πολιτισμός είναι ένα εργαλείο. Έχουμε διαφορετικές αφετηρίες λοιπόν, που με τρόπο λογικό θα πρέπει να συγκεραστούν και να συγχωνευτούν. Και στη συνεργασία με την κυρία Κώστα νομίζω τα καταφέραμε. Και επίσης αν συμπεριλάβουμε τον πολιτισμό και τις αξίες που συνδέονται με αυτόν, θα μπορέσουμε να βρούμε και συμβιβασμούς και μετριοπαθείς τάσει. γενικότερα, να δρούμε ειρηνευτικά και θα πρέπει να καταλάβουμε ότι η ιστορία και ο πολιτισμός παίζουν σημαντικό ρόλο. Εγώ όταν πηγαίνω στο εξωτερικό πάντα προετοιμάζομαι. Διαβάζω την ιστορία και τον πολιτισμό της κάθε χώρας που επισκέπτομαι. Και αυτό είναι πολύ βαθύτερο από τα οικονομικά στοιχεία που ή αλλάζουν. Οπότε καταλαβαίνετε ότι και αυτό είναι σημαντικό που θα πρέπει να λαμβάνετε υπόψη. Αλλά θα πρέπει και τα κράτη-μέλη να μας ακολουθήσουν. Ο πολιτισμός δεν είναι ευρωπαϊκή αρμοδιότητα, είναι αρμοδιότητα των κρατών μελών. Τα πολιτιστικά θέματα είναι στην κατηγορία 3 της ε, ε, συνθήκης Λισαβόνας. Δηλαδή εμείς παίζουμε ένα ρόλο μόνο υποστηρικτικό το πολύ πολύ. Άρα τα κράτη-μέλη θα πρέπει να ενδιαφερθούν να συμμετέχουν. Και πιστεύουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να βοηθήσει έτσι ώστε τα κράτη-μέλη σε συνεννόηση μεταξύ τους να παρουσιάσουν και να προβάλλουν και εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης την πολιτιστική τους κληρονομιά και την πολιτιστική τους πολυφωνία. Έτσι μπορούμε και να παρουσιάζουμε και να προβάλλουμε την ταυτότητά μας την ίδια και την ταυτότητα των κρατών μελών και να πούμε ότι είναι προστιθέμενη αξία και υπεραξία της Ευρώπης. Επιχειρησιακά δηλαδή να χρησιμοποιούμε τον πολιτισμό ε, και στη συνεργασία μας αλλά και για την προβολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και να αναπτύσσουμε ένα επιπλέον στοιχείο πολιτικής χρήσιμο για τη δράση μας. Και επαναλαμβάνω ότι είχαμε καλή συνεργασία με την κυρία Κώστα και διαφορές έχουμε ακόμα σε αυτή τη συμβαστική τροπολογία περιθμών 2 μεταξύ των διαφόρων ομάδων. Θα φύγω τώρα, αλλά με περιμένω στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για ένα πολύ πολιτιστικό θέμα. Δηλαδή, με ποιον τρόπο το Ινστιτούτο της Φλωρεντίας, το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο μπορεί να αναπτυχθεί ως Ευρωπαϊκή Διπλωματική Σχολή με διεθνή ακτινοβολία. και επειδή έχουν έρθει εκπρόσωποι ε, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή μου ζήτησαν να είμαι παρόν στην αρχή της συζήτησης για να τους υποστηρίξω, για να προωθήσουμε και αυτό το εγχείρημα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε κύριε Μπροκ και τώρα ο λόγος στην κυρία Κώστα. Ε, buonasera a tutti, mi scuso per σας ευχαριστώ, συγγνώμη για την καθυστέρηση. Μετά από τον κύριο Μπρόκ, ο οποίος υπογράμμισε τα πιο βασικά στοιχεία τα οποία έχουν έρθει στην επιφάνεια μετά από τις συζητήσεις που έγιναν, να πω πάρα πολύ σύντομα ότι υπό το φως των τροπολογιών που έχουν κατατεθεί αποδεικνύεται το ενδιαφέρον του κειμένου Συνολικά οι τροπολογίες αυτό το οποίο ζητούν είναι να ακολουθηθούν ορισμένοι προσανατολισμοί τους οποίους προσπαθήσαμε με τον συνεισηγητή να ορίσουμε ε, και εκεί ακριβώς προσαρμόσαμε τις προτάσεις για αλλαγές ε, μέσω των συμβιβαστικών. Εμείς υπογραμμίζουμε τα πλαίσια στο εσωτερικό των οποίων ε, θα γίνει η συζήτηση και με την Επιτροπή, το πλαίσιο δηλαδή του πολιτισμού στον τομέα των διεθνών σχέσεων που θα πρέπει να χαρακτηρίζονται πάντα από μια πολιτιστική διάσταση και ακόμα και η αναφορά στην εκπαίδευση και την έρευνα είναι βασικά στοιχεία για την αναζήτηση ενός πραγματικού στρατηγικού ρόλου και δίδοντας το μήνυμα αν θέλετε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει να αναλάβει έναν σημαντικότατο ρόλο πρωταγωνιστή στον τομέα της ειρήνευσης, του διαπολιτιστικού διαλόγου, του διαθρησκευτικού διαλόγου και των πολιτιστικών σχέσεων που όπως είπανε πολλοί από τους καταθέτοντες της τροπολογίες θα πρέπει να διεξάγονται πάντα σε μια υποχρέωση έτσι ώστε όλες οι διεθνείς συμφωνίες και όλες οι συζητήσεις οι οποίες γίνονται σαν παράδειγμα με τη ΣΑΚΕ να λαμβάνουν υπόψη και την διαπολιτισμική διάσταση. Νομίζω λοιπόν ότι το πνεύμα αυτό χαρακτηρίζει πάρα πολλές από τις τροπολογίες, το λάβαμε υπόψη μας στις συμβιβαστικές, καταθέτουμε 20 συμβιβαστικές οι οποίες ε, εκπροσωπούν ε, δεκάδες τροπολογίες, θα θέλαμε να ενσωματώσουμε και τις υπόλοιπες όπου αυτό είναι εφικτό. Προτείνουμε λοιπόν συγκεκριμένους στόχους στον τομέα της διακυβέρνησης, ε, της αντιμετώπισης people to people. Επίσης ε, εμείς ε, δεχόμαστε τις τροπολογίες οι οποίες δείχνουν την εσωτερική αξία του πολιτισμού, το λεγόμενο soft power, την ήπια δύναμη, στα πλαίσια μιας υψηλότερης ακόμα επικουρικότητας, Πρόκειται για μια πλατφόρμα η οποία εκπροσωπείται από τις τροπολογίες που ζητούν να καταστεί ο πολιτισμός σημείο αναφοράς Επίσης η σημασία την οποία έχουν τα διαπολιτισμικά δίκτυα και οι εμπλεκόμενοι στα δίκτυα αυτά όπως η UNESCO, το Συμβούλιο της Ευρώπης, και μια ολόκληρη σειρά από οργανισμούς. Ένα άλλο σημαντικό θέμα στο οποίο έγινε αναφορά είναι ο πολιτισμός ε, ε, στα πλαίσια του διαφρομένου διαλόγου για την διακυβέρνηση. Δηλαδή, θα πρέπει εδώ να λάβουμε υπόψη μας τους μηχανισμούς που εκπροσωπούν τους δημιουργούς αλλά και τα δίκτυα διανομής, ο ρόλος της κοινωνίας των πολιτών στα πλαίσια της εμπλοκής των ε, πολιτιστικών πρωταγωνιστών αν θέλετε, ενίσχυση της διεθνούς διάστασης των ε, προγραμμάτων που είναι ήδη εν λειτουργία και ταυτόχρονα ενίσχυση του ρόλου των δημιουργικών και πολιτισμικών βιομηχανιών στον τομέα της κοινωνικής και ανάπτυξης. Πρέπει λοιπόν να δούμε και η πολιτιστική κληρονομιά πώς ε, μπορεί να γίνει αντικείμενο έκφρασης και μέσα από έναν ταχύτατο μηχανισμό δράσης, κάτι το οποίο συμβαίνει ε, και μέσα από τη δράση της UNESCO σε διάφορες χώρες η πολιτιστική διάσταση θα πρέπει, ή μάλλον οι παραβάσεις εις βάρος του πολιτισμού και τα εγκλήματα εις βάρος του πολιτισμού θα πρέπει να θεωρούνται εγκλήματα εις βάρος της ανθρωπότητας και θα πρέπει να εκφράσουμε την ανησυχία μας για μία μορφή διακυβέρνησης με συγκεκριμένους τρόπους και συγκεκριμένες χρονικές προθεσμίες. Υπάρχουν κάποια πολυμερή πολυετή προγράμματα στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Φόρουμ για τον Πολιτισμό και των ημερίδων ε, για την πολιτιστική ανάπτυξη πολιτική γειτονίας και πολιτισμός και με την Ανατολή και με τον Νότο της Ευρώπης. Και τέλος αυτό το οποίο έχει σημασία είναι να υπογραμμίσουμε τις νέα, τη νέα γενιά, τις νέες γενιές, στα πλαίσια ενός προγράμματος κινητικότητας των νέων καλλιτεχνών και επίσης να γίνουν και κάποιες επιπλέον αναφορές που προτείνονται από αρκετού συναδέλφους να καταλήξουμε σε μία ποιότητα, σε μία χάρτα ποιότητας, σε κάποιους δείκτες και σε κάποια δεδομένα τα οποία θα διευκολύνουν την αξιολόγηση του πολιτισμού και αυτό θα καλύπτει και τον πολιτισμό των μεταναστών και των μειονοτήτων. Είναι σημαντικό ότι το 2018 που θα είναι το έτος για την, για την πολιτιστική κληρονομιά θα είναι και το έτος εκκίνησης αυτής της στρατηγικής. Και τέλος ξανά λέει η Πρόεδρος, να μπορέσουμε να στρέψουμε σωστά την προσοχή μας στις εμπορικές ε, σχέσεις και του τρόπου με τον οποίο άπτονται ε, της πολιτιστικής κληρονομιάς ε, και της εισαγωγής των πολιτιστικών αγαθών σε περιπτώσεις συγκρούσεων, πολέμων κτλ. Όλα αυτά θα πρέπει λοιπόν να ληφθούν υπόψη. Νομίζω ότι θα κάνουμε για κάποιες άλλες συμβιβαστικές για το σύνολο των 320 τροπολογιών. Στις 30 Μαΐου θα γίνει η ψηφοφορία και μέχρι τότε ελπίζω να δουλέψουμε πολύ καλά με τους χιώδεις. Σας ευχαριστώ πολύ. για το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. ο κύριος Ντρογεύσκη. Καταρχάς, σχετικά με τις συμβιβαστικές. Νομίζω ότι οι συμβιβαστικές είναι χρήσιμες και συμπεριλαμβάνουν την πλειοψηφία των τροπολογιών και γι' αυτό δεν θα πρέπει να αλλάξουν άλλο. Όπως είπε και ο κύριος Μπρόκ στην αρχή, υπάρχουν κάποιες διαφορές μεταξύ μας σαν για τις δύο τροπολογίες από αυτές νομίζω ότι δεν πρέπει να βάζουμε ονόματα τώρα γιατί αν βάλουμε ας πούμε το όνομα του Λάιμπνιτς θα πρέπει να βάλουμε και το Βολτέρ θα πρέπει να βάλουμε και άλλους. Αν βάλουμε το όνομα του Ισλάμ είναι σαφές ότι θα πρέπει να βάλουμε και άλλους πολιτισμούς άλλων χωρών που έχουν επηρεάσει μεταξύ των οποίων και τον Ιαπωνικό πολιτισμό που έχει επηρεάσει τον Ευρωπαϊκό πολιτισμό στον τομέα της γαστρονομίας. Jeżeli dziś tym dokumentem zwracamy uwagę na istotę kultury, Λοιπόν, θα πρέπει να συγκεντρώσουμε την προσοχή, μας, την προσοχή μας στην ουσία του πολιτισμού, στον τομέα του απτού πολιτισμού, αλλά και του πνευματικού πολιτισμού της Ευρώπης. Εμείς λέμε ότι ο πολιτισμός είναι ένα στοιχείο αξίας που πρέπει να χρησιμοποιείται και στη διπλωματία. Και αυτό είναι ένα καλό βήμα προς τα εμπρός. Να μην ξεχνάμε όμως ότι στα πλαίσια της στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης ο πολιτισμός προάγεται μέσω της προαγωγής, ε, μέσω των τρόπων που επιλέγουν τα κράτη-μέλη ξεχωριστά. Οπότε αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να συνδυάσουμε. Θα πρέπει επίσης να στηρίξουμε τις συμβιβαστικές και να μην προσπαθήσουμε να πλουτίσουμε ακόμα περισσότερο το έγγραφο. Σας ευχαριστώ πολύ. Η επόμενη ομιλήτρια, η κυρία Χιμένες. Κυρία σας. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τη Σίλβια Κώστα για τη δουλειά της στην έκθεση για τη στρατηγική της Ένωσης για τις ε, διεθνείς πολιτιστικές οργανώσεις και για το γεγονός ότι συμπεριέλαβα και κάποιες από τις προτάσεις μου μέσω τροπολογιών ε, στις συμβαστικές της ε, τροπολογίες. Η έκθεση αυτή περιλαμβάνει τις ιδέες και τις αξίες ε, για τον πολιτισμό που είναι κοινέ για όλους μας. Υπάρχει δυνατότητα να γεφυρώσουμε λοιπόν τις σχέσεις ατόμων πάσας προέλευσης και αυτό φυσικά είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί μπορεί να βοηθήσει και την εξωτερική πολιτική της Ένωσης. Θα ήθελα να σταθώ σε κάποια σημεία ε, από τη συζήτηση που είχαμε στην πρώτη συνεδρίαση των σχεδόν εισηγητών. Θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικός ο διάλογος μεταξύ πολιτισμών και θρησκειών, αλλά ταυτόχρονα ο διάλογος αυτός πρέπει να περιλαμβάνει και ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν κάποια θρησκευτική πεποίθηση, ανθρωπιστές, ανθρώπους οι οποίοι έχουν ελεύθερη σκέψη και δεν ε, είναι πιστοί ε, και εκπροσωπούν ένα πολύ σημαντικό ποσοστό του παγκόσμιου πληθυσμού. Αυτοί οι άνθρωποι ζουν ε, παντού και σε χώρες όπου κυριαρχεί ε, η μουσουλμανική θρησκεία. Θεωρώ λοιπόν ότι θα πρέπει να αναγνωρίσουμε αυτούς τους ανθρώπους, ιδέως αν θέλουμε να ε, συμπεριλάβουμε τις ανθρωπιστικές αξίες της ελευθερίας συνείδησης ε, που είναι πάρα πολύ σημαντικές και αποτελούν θεμέλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η διάρθρωση αυτής της έκθεσης θέλει να βοηθήσει την πολιτιστική συνεργασία μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και χωρών εταίρων και θα πρέπει να βασίζεται στη διατήρηση της ειρήνης και στη μείωση των συγκρούσεων μέσω του σεβασμού του κράτους δικαίου. Η ελευθερία έκφραση και τα ανθρώπινα δικαιώματα προέχουν. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Μιγιάν Μον. Μίλαν Μον. Έχετε το λόγο. Συγγνώμη, Μιλούσα για τις συμβαστικές τροπολογίες, γιατί ε, μου είπαν ότι έχουμε αποδεχτεί κάποιες τροπολογίες, αλλά εγώ δεν είχα την τύχη να μάθω για αυτά τα κείμενα. Μετά λοιπόν από αυτή τη διευκρίνηση θα ήθελα να ευχαριστήσω και πάλι τη Σίλβια Κώστα και τον Έλμαρ Μπρόκ για την έκθεσή τους. Οι πολιτιστικές σχέσεις είναι πάρα πολύ σημαντικές ε, για την Ευρώπη στο διεθνές ε, προσκήνιο και η Ευρώπη και τα κράτη-μέλη είναι δυνητικά πολιτιστικές δυνάμεις. Επομένως, αν το δούμε ε, ως ένα εργαλείο τον πολιτισμό, κατά πάσα πιθανότητα θα πρέπει να μπορούμε να τον εκμεταλλευτούμε και να τον εκμεταλλευτούμε και καταλήλως για μια ε, οντότητα όπως είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση, το να έχει ε, σχέσεις πολιτιστικής φύσεως έχει κάποια ε, σημασία γιατί μπορούμε να συντονιστούμε με τα κράτη-μέλη και να μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε τον πολιτισμό ως διεθνές εργαλείο. Θα ήθελα να σταθώ εδώ στις λεγόμενες πολιτιστικές διαδρομές. Είναι κάτι το οποίο ξεκίνησε πριν από 30 χρόνια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πριν από 30 χρόνια είχαμε λοιπόν τη διαδρομή του Σαντ και ε, οι πολιτιστικές διαδρομές ε, δεσμεύουν αρκετά κράτη-μέλη. Έχουμε ήδη 32 διαδρομές ε, με χώρες της ανατολικής και νότιας γειτονίας. Πρόκειται για κοινού χώρους, κοινέ ρίζες ε, και ο πολιτισμός είναι ένας θετικός δεσμός, ε, δεν χωρίζει αλλά ενώνει για να μπορέσουμε να κάνουμε διάλογο και όχι μάχες και να συνεννοηθούμε. Και θεωρούμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό και θα πρέπει να συνεχίσει να το υποστηρίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση και θα ήθελα να τονίσω εδώ και με αυτό ολοκληρώνω ότι αυτές οι διαδρομές δεν θα πρέπει να μείνουν μόνο στις ε, χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά θα πρέπει να επεκταθούν και σε υποψήφιες χώρες και σε χώρες της πολιτικής γειτονίας. Θα ήθελα να πω στην κυρία Κώστα και στον κύριο Μπρόκ που μας εγκατέλειψε να δουν με θετικό ε, πνεύμα την ε, τροπολογία 310 που θέλει να ενισχύσει τους δεσμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης με αυτό το πολύ σημαντικό πρόγραμμα του Συμβουλίου της Ευρώπης. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Δεν έχουμε άλλον που να έχει ζητήσει το λόγο, οπότε η κυρία Κώστα και πάλι.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 Ευχαριστώ τους συναδέλφους και να ευχαριστήσω και τον συνάδελφο Μπρόκ και τους και οδησηγητές γιατί έχουμε κάνει αρκετή δουλειά στις συμβαστικές τροπάσεις και θα ήθελα να καθησυχάσω και τον κύριο Μιγιαμόν ότι έχουμε την ίδια ανησυχία για αυτές τις διαδρομές και το είχαμε προβλέψει αλλά το ενισχύσαμε κιόλα διότι είναι και μια στρατηγική πιο στενών σχέσεων με τη Συμβούλιο της Ευρώπης. Σίγουρα λοιπόν απαντάμε καταφατικά σε αυτή την πρόταση. Να απαντήσω και στους συναδέλφους που μίλησαν προηγουμένως Σίγουρα κύριε Σδρογεύσκη και εγώ θεωρώ ότι πρέπει να βλέπουμε μπροστά και να δούμε τι είναι αυτά τα οποία μας ενώνουν και να έχουμε και ε, κάτι συγκεκριμένο πλέον για μια διεθνή ε, πολιτιστική πολιτική σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Το είπα βέβαια και λαμβάνοντας υπόψη την επικουρικότητα. Αναφερόμαστε στην πλατφόρμα της πολιτιστικής διάστασης που θα περιλαμβάνει και εθνικά πολιτιστικά ιδρύματα και άλλα πολύ σημαντικά ιδρύματα. Αλλά εγώ θεωρώ ότι ε, το θετικό βήμα προς το κατεύθυνση είναι, όπως προβλέπει και το άρθρο 167 των συνθήκων, να ε, τα αντικαταστήσουμε με πολιτικές οι οποίες θα προβάλλουν καλύτερα και θα ενισχύουν την Ευρωπαϊκή Ένωση και θα ενισχύσουν και τη συνεργασία σε τρίτες χώρες ε, των πρωτοβουλειών που λαμβάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε πολιτιστικό επίπεδο και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρέπει να έχουμε λοιπόν κοινά προγράμματα αλλά και κοινέ ρίζες. Για να απαντήσω στην ε, συνάδελφο Χιμένεθ, που είναι εκεί στο βάθος. Θα ήθελα να ε, πω ότι σαφώς ε, αντιλαμβανόμαστε την ανησυχία σας. Όταν αναφερόμαστε σε διαπολιτιστικά και διαθεσκευτικά, κατά την άποψή μου, συγγνώμη δεν μπορώ και να γυρνάω πίσω, σημαίνει και όλους εκείνους που δεν είναι πιστοί. είμαστε ανοιχτοί σε όλες τις φιλοσοφίες και σε όλους τους πολιτισμούς. Θεωρώ ότι αυτό είναι αυτονόητο, αλλά αν θέλετε να διασκεδάσουμε και την ανησυχία της, νομίζω ότι μπορούμε να βρούμε μια λύση. Ε, αυτή τη στιγμή υπάρχει μια πολύ μεγάλη πρόκληση που αφορά το διαθρησκευτικό διάλογο που είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό πολύτιμο αγαθό για όλους και για αυτούς που δεν πιστεύουν διότι υπάρχει έτσι δυνατότητα να εφαρμόσουμε πολιτικές ειρήνης και ενίσχυσης των κοινών αρχών πέραν των θρησκειών. Και νομίζω ότι η συνάντηση που έγινε στην Αίγυπτο αυτές τις μέρες του Πάπα Φραγκίσκου με άλλες ε, εκπροσώπους άλλων θρησκειών ε, δείχνει και την υποχρέωση που έχουν οι ίδιες οι θρησκείες ε, να προωθήσουν αυτό τον ε, διαπολιτισμικό και διαθρησκευτικό διάλογο. Αλλά αυτό σημαίνει και άνοιγμα προς όλους και σε προσωπικά πιστεύω και σε διαφορετικούς πολιτισμούς και πολιτιστικές ρίζες και σε εθνικό επίπεδο. Όσον αφορά το στοιχείο το οποίο προβάλλετε και εσείς, συμφωνώ και το ξέρετε και στις συμβαστικέ προτάσεις, ε, διότι συμμετείχατε και στις συνεδρίες των σκεδών εισηγητών, προσπαθήσαμε να το συμπεριλάβουμε. Τη διατήρηση της ειρήνης, ε, της διακοπής των σειράξεων και το γεγονός ότι θα πρέπει να ε, υπάρχει και συνδυασμός με τις θεμελιώδεις ανθρώπινες αξίες και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Αυτά, ευχαριστώ πολύ. Νομίζω με τον συνάδελφο Μπρόκ θα διαφερθούμε και με όλα αυτά και θεωρώ ότι ήταν πολύ σημαντικό να μπορέσουμε να συζητήσουμε από κοινού αυτέ τι προτάσει. Ευχαριστώ πολύ. Και Εγώ σας ευχαριστώ. Και τώρα... Μπορούμε να κηρύξουμε τη λήξη της κοινή συνεδρίασης Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας. Καλό σας απόγευμα. Ευχαριστώ τα μέλη της Επιτροπής Πολιτισμού σε αυτή τη κοινή συνεδρίαση. Ε, λέει ο πρόεδρος της Επιτροπής ΑΦΕΤ, ο Προεδρεύων, παρακαλώ υποχωρήστε ησύχως, γιατί εμείς στην ΑΦΕΤ έχουμε τώρα ψηφοφορία ως επόμενο θέμα που αρχίζει αμέσως. Λοιπόν, έχετε 30 δεύτερα για να βγείτε και ακολουθεί ψηφοφορία.